Ε, Όντω υπάρχουν κίνδυνοι, δεν ε, έχουμε έτοιμε λύσει, αλλά πρόκειται για ένα βήμα το οποίο μα έχει κάνει περήφανο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, λέει Πρόεδρο. Πρώτα-πρώτα να με συγχωρούν οι δύο συνάδελφοι που τους διέκοψα εν τη ροή της ομιλίας τους αλλά μόλις ε, αντικατέστησα τον προηγούμενο αντιπρόεδρο μου είπαν θα πρέπει να προβούμε σε κάποια ανακοίνωση παρακαλώ προσέξτε με ο κύριος Κριστόφ Μπεσί με ενημέρωσε ότι παρετείται ως Ευρωβουλευτής και απόφαση αυτή ανατρέχει σε σχέση με την 1η Πρώτη 2011. Δυνάμει. Τη διατάξεω 4, πρώτη παραγράφου, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η θέση χειρεύει από εκείνη ημερομηνία. Οι δέκα γαλλικέ αρχέ μα είπαν ότι ο αντικαταστάτη, η αντικαταστάτη του κ. Κριστόφ είναι η κυρία Νιέ Λεμπρέ και σύμφωνα με την διάταξη 4 παράγραφο 1, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ανέλαβε τα καθηκοντά τη από την αντίστοιχη ημερομηνία 1η 1η 2011 και σύμφωνα με την διάταξη 3 παράγραφο 2, μέχρι ότου πιστοποιηθεί ο διορισμό τη ε, και διαπίστευσή τη και έχουν, δεν υπάρχουν άλλες ενστάσεις θα λάβει τη θέση της, θα έχει όλα τα προνόμια, ασυλίες, όμως θα πρέπει να υπογράψει τη γνωστή δήλωση ότι δηλαδή δεν κατέχει κάποια θέση συμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και, ευχόμαι θέση στην Γεωργία συνάδελφο καλή επιτυχία. Και τώρα επιστροφή στη συζήτησή μας. Ο επόμενος ομιλητής. Η κυρία Ζολή, εκ μέρους της Επιτροπής Αναπτύξεως για να Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι συμφωνίε εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καμερούν ή Κονγκό πρέπει να αποτελέσουν καταρχήν καλή είδηση, καλά νέα για τους λαούς τους, τους λαούς των χωρών αυτών, αλλά και για τη βιοπικιλότητα. Είναι όμως ένα στάδιο, μια μακρά διαδικασία την οποία το Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει με επαγρύπνηση ναι, θέλουμε να έχουμε εμπόριο ξυλίας διαφανές, εύρυθμο, που θα αποβαίνει σ' των τοπικών πληθυσμών και όχι κάποιων κατά το μάλλον ή των νόμιμων ομήλων και γι' αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να τύχουν πλήρους σεβασμού τα δικαιώματα των πληθυσμών στην περιοχή αυτή και το δικαίωμα για διαβούλευση. Θα πρέπει η εταιρική σχέση να ενισχύει τη συμμετοχή των παραγόντων αυτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τη θέσπιση μιας ουσιαστικής διακυβέρνησης για τα δάση. Δεν πρέπει αυτές οι συμφωνίες να αποτελέσουν πρόσχημα για διαιώνιση της ε, ε, καταστροφής των δασών και του σφετερισμού των πόρων τους, αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν ένα εργαλείο ανάπτυξης των κρατών. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και πρώτον εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Φιέλνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την ε, συζήτηση που έχουμε σήμερα για τις συμφωνίες με το Καμερούν και το Κονγκόν. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, είναι πολύ σημαντική η συμφωνία, συμφωνίες και γι' αυτό τις χαιρετίζω. Η δασπονία, ο δασικό τομέα έχει πολύ μεγάλη, σημασία, πολύ μεγάλη σημασία και οικονομική αλλά και κοινωνική. Έτσι λοιπόν η παράνομη, η λαθρέα υλοτομία έχει τεράστια σημασία και επιπτώσεις που φτάνουν μέχρι τη φτώχεια, τη διαφθορά, τους πολέμους ακόμη που βλέπουμε να ξεσπούν μεταξύ των παράνομων αυτών ομάδων ξυλοτομίας. Και με χαρά βλέπω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση στην υπόθεση αυτή. Στόχος μας είναι βέβαια το ελεύθερο εμπόριο και γι' αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα κανόνες που θα επιτρέπουν την, την πάταξη της διαφθοράς. Και βεβαίως θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε με τα συμπτώματα του φαινομένου αυτού μέσα από τις συμφωνίες αυτές. Θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να δούμε τη σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών και με περισσότερα κράτη, διότι Εάν δεν παταχθεί αυτής, αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς, δεν θα έχει αυτή η προσπάθεια κανένα νόημα. Δεν θα έχουμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ε, εισαγωγών παράνομης ξυλίας ή ξυλίας που έχει υλοτομηθεί παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σουηδία Φερρυπίνη, η οποία έχει μεγάλη παραγωγή ξυλίας, αλλά εισάγει και από φτωχότερα από ότι εμείς κράτη πάλι είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους ίδιους κανόνες που τηρούν οι άλλοι και αυτό για να έχουμε την ευκαιρία να πατάξουμε όλοι μαζί την διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσούτας εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία εταιρική σχέση με τις χώρες εξαγωγούς ξυλίας. Ενώ πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να εκπονήσουμε μία δομή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων ώστε να εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών και να βελτιώσουμε το πλαίσιο της διακυβέρνηση των δασών ώστε να αποφευθεί στο μέτρο του δυνατού η διαφθορά. Η εμπλοκή τη της κοινωνίας των πολιτών στη συμφωνία, στη διαπραγμάτευση μάλλον της συμφωνίας με το Καμερούν είναι ένα θετικό στοιχείο. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να συνεχιστεί ο διάλογος σε όλες τις συνυπογράφησες χώρες. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια βιομηχανία βιώσιμη το, για την εξηλία και να αποφευθεί η αποψήλωση αλλά και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις χώρες αυτές. Να τονίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να σεβαστούν τη, της ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την δασική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ντέβις, λεπτό. Μιλούμε για αυτές τις τελευταίες εταιρικές συμφωνίες και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία λόγια. Πολύ συμπαθήκα και λέμε ότι δεν θέλουμε να τους επιβάλλουμε τίποτα τις, ε, αυτές τις χώρες. Απλώς θέλουμε να τις βοηθήσουμε και έτσι να μπορέσουν να προχωρήσουν προς κοινούς στόχους. Όμως, όμως η ομή πραγματικότητα, δηλαδή το τεράστιο μέγεθος της χώρας αυτής δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα και το μέγεθος, μόνο και μόνο το μέγεθος αυτή τη χώρα, ξέρετε ότι η είναι σχεδόν αυτό τη Ευρώπη, οπότε η διακυβέρνηση τη χώρα είναι κάτι το απίστευτο, αδύνατον. Και οπότε γι' αυτό λέμε ότι η διεθνή ε, διαφάνεια είναι κορυφαία στη διαφθορά. Οπότε το προσωπικό το οποίο έχουν στη διάθεσή μα ε, δεν μπορεί να βοηθήσει τόσο να πετύχουν του σχολείου. Γιατί πρόκειται για μια χούφτα ανθρώπου. Τα κέρδη από την παράνομη λοτομία είναι τεράστια. Είναι ο, καμία σχέση με αυτό που του δίνουμε εμεί. Κίνα, α πούμε, είναι αγορέ που πληρώνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμεί. Αυτοί πληρώνουν για να πάρουν το ξυλία και εμεί για να διατηρηθεί και έχουμε τόσα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι εθελοντικές εταιρικέ σχέσεις προσκούν σε αυτές τις δυσκολίες. Πώς μπορεί να μας καθησυχάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κάνει ό,τι γίνεται ούτω ώστε να υπάρξουν φιλόδοξοι στόχοι και εμείς να θεωρήσουμε ότι θα έχουν αίσιο πέρα σε αυτές τις συμφωνίες. Η πρόταση ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα για τους φιλεύθερους δημοκράτες. κύριε Ρόσπαχ. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα δάση είναι η μας του πλανήτη και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα προστατεύσουμε. Συχνά πρόκειται για πόρους που τους υπερεκμεταλλευόμαστε. Εμείς έχουμε τη συνήθεια να εισάγουμε τροπική ξυλία, ωστόσο ε, δεν σκεφτόμαστε ότι προέρχεται από χώρες ε, που είναι διεφθαρμένες και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ε, διαφθορά εκεί. Έτσι βλάπτεται η βιοπικιλότητα. Πρόκειται για φυτά, ζώα που μας βοηθούν να προστατευτούμε από τις κλιματικές αλλαγές. Δεν υπάρχει ανελαλλακτική από αυτά τα τροπικά δάση και η Ευρώπη θα πρέπει να δεσμευτεί υπέρ της μείωσης ε, της εκμετάλλευσης των δασών αυτών. Ωραία και καλά είναι να έχουμε εξωτικό ξύλο στο παρκέ μας στην Ευρώπη, όμως όταν μιλάμε για εμπορία τροπικό, τροπικής ξυλίας θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συμφωνία, να υπάρχουν όροι, συνθήκες ξεκάθαρες για την ε, εισαγωγή τέτοιες τροπικής ξυλίας. Εγώ δυστυχώ δεν είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να καταργήσουμε την παράνομη υλοτόμηση των δασών στο Κονγκό ή στο Καμερούν. Πάντω είναι καλύτερο να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία παρά να μην υπάρχει καθόλου συμφωνία και γι' αυτό την υποστηρίζω. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερε ε, μελλοντικέ πρωτοβουλίε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε προβληματικέ χώρε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ και Σμόλτσερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι συμφωνητερικέ ε, σχέσεις τη στη, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Καμερούν έρχεται την κατάλληλη στιγμή πιστεύω και μάλιστα την Ευρωπαϊκή, το, Διεθνέ Διεθνές Έτος Προστασίας των Δασών. Βέβαια το πρόβλημα της διαφθορά του Καμερούν είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο και ασφαλώς γνωρίζει η κυβέρνηση. Η πρόεδρος Λέω ότι δεν ακούγεται η διερμηνία. Εάν θέλετε να ξαναρχίσετε κύριε Μιόλτσερ, μπορείτε να ε, αρχίσετε από την αρχή την ομιλία σας γιατί σας άκουσαν όλοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση για τα θέματα τη διαχείριση των δασών με το Καμερούν ε, είναι πολύ σημαντική και σε κατάλληλη χρονική στιγμή, δηλαδή ε, το έτος Προστασία των δασών έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα διαφθορά στο Καμερούν και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν την κυβέρνηση ότι είναι εν γνώση της εγκληματικής δραστηριότητας των ομίλων ε, υλοτομίας και οι οποίοι ελέγχουν ε, μέχρι τρία τέταρτα των εξαγωγών ξυλίας ε, από το Καμερούν προς τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπουμε επίσης ότι χάνεται η τεχνογνωσία ε, από τον λαό του Καμερούν και η προστασία των τροπικών δασών δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και στην Ευρώπη να έχουμε αντίστοιχη προστασία και ορθή διαχείριση των ε, δασών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τη διπλή σας επίδοση. Ευχαριστώ. Κύριο Σκάτσμαρεκ τώρα για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν από ένα μήνα, μαζί με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης, επισκέφθηκα την ε, ε, το Κονγκό, όπου είχα και την ευκαιρία να συζητήσω με εκπροσώπους των εθνικών αρχών αλλά και των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η βιομηχανία της ξυλίας είναι ένας ε, πολύ σημαντικός παράγων τομέας οικονομικός στο Κονγκό. Είναι η δεύτερη σε έσοδα κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας και μην ξεχνάμε ότι για το πετρέλαιο που είναι η πρώτη πηγή εισόδων στο Κονγκό, έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, ελάχιστη διαφάνεια, δεν ξέρουμε πώς γίνεται η εξόριξή του. Το ίδιο λοιπόν βλέπουμε ως φαινόμενο συμβαίνει και στην ε, περίπτωση της ξυλίας. Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει ικανοποιητικά λοιπόν και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ενισχύσει την νόμιμη διακίνηση ξυλίας. Ελπίζουμε δε να ε, δώσει έμπνευση και να επεκταθεί η νόμιμη υλοτομία και στις υπόλοιπες χώρες για να μην ε, βρουν διαφορετικούς διάβλους ε, τα δίκτυα παράνομης υλοτομίας τα οποία βέβαια ξέρουμε ότι δρούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι αυτό. Το σύστημα λοιπόν το οποίο προτείνεται θα πρέπει να γίνει στο δυνατόν πιο αξιόπιστο και ευρύ έτσι ώστε να παταχθεί σταδιακά αλλά αποφασιστικά η παράνομη υλοτομία. Η ανάπτυξη λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσει κατά τρόπο ουσιαστικό στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής οικονομική ανάπτυξη και βιομηχανία τροφίμων καθώς και υλοτομία ε, διαφανής και βιώσιμη. Ευχαριστώ κύριο Στασέλη, ένα μισή λεπτό. Επίτροπε, καταρχήν τα συγχαρητήριά μου για την ε, ολοκληρώση στην ουσία των ε, διαπραγματεύσεων για τις δύο αυτές συμφωνίες, αλλά και η ανησυχία μου γιατί έχουν παγώσει διαδικασίες με την διαπραγμάτευση τη της διαδικασίας με την Ινδονησία και τη Μαλαισία. Επίτροπε, ως Επιτροπή έχετε στα χέρια σας ένα σημαντικό εργαλείο, τον κανονισμό για τη ξυλία αυτό το εργαλείο εξαιρεί τις χώρες που έχουμε συμφωνία flegt από τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός. είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δώσουμε νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις γιατί χρειαζόμαστε ε, να ολοκληρώσουμε συμφωνίες flegt με όλες τις χώρες που έχουν σημαντικά τροπικά δάση είτε στην ασία είτε στην λατινική αμερική αλλά και του μεγάλους μεταπράτες της ξυλίας είτε αυτή είναι το βιετνάμ η Καμπόζη, το Λάο, η κίνα και τόσε άλλε χώρες. επίσης αυτές οι χώρες κάνουν το δικό τους κομμάτι προχωράνε στις δικές τους διαδικασίες για να εξυγχρονιστούν να μπορούν να παρακολουθούν ε, την ε, νόμιμη ε, υλοτόμηση. το ερώτημα είναι εμείς κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. τα κράτη μέλη τα 27 κράτη μέλη παίρνουν τις κανονιστικές αποφάσεις προκειμένου αναφορικά με τις εισαγωγή ξυλίας από χώρες ΦΛΕΚΤ. και τέλος για το κανονισμό της ξυλίας ε, απαιτούνται μια σειρά από delegated acts. Ε, έχουμε δύο χρόνια μπροστά μα για την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού. Χρειάζεται η Επιτροπή πραγματικά να επισπεύσει τι διαδικασίε, να προχωρήσουμε σε αυτά τα delegated acts, να γνωρίζουν οι χώρε τι λεπτομέρειε στι οποίε πρέπει να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στο ε, διαδικασία Catch the Eye. Δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλους όσους το ζήτησαν. Πρώτος ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ πιο σημαντικό το θέμα από τη δημοσιότητα που θα λάβει, όμως τα σκάνδαλα Ε, είναι πολύ μεγαλύτερα. Ε, μεγάλες ε, πολυεθνικές, λέμαργες κυβερνήσεις είναι αυτές που καταστρέφουν τα πάντα. Ελπίζω πως αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί γιατί διαφορετικά δεν θα αξίζει τον κόπο που κάναμε. Και ελπίζω πως και τα κράτη θα συμμετέχουν, θα εμπλακούν. Ιδιαίτερα φέρουμε στη συμφωνία με το Μερκοσούρ ε, γιατί πολλοί κόσμος ε, συνομίζει πως ε, εμείς ενθαρρύνουμε την αποψήλωση των δασών για τα βιοκαύσιμα. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εκμετάλλευση, παράνομη εκμετάλλευση ξυλίας στις χώρες κεντρικής Αφρικής όπως το Καμερούν και το Κονγκό αποτελεί απειλή στους πόρους ε, από τους οποίους εξαρτώνται οι τοπικές ε, κοινότητες και οι αυτόχθονες ε, πληθυσμοί είναι μια μεγάλη απειλή για τη βιοπικιλότητα. Μεγάλη σημασία θα επίσης παίζει για την ρύθμιση των βιοχημικών κύκλων. Η διασυντήρηση λοιπόν των τροπικών δασών σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να δοθεί με μέσω τη ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται μόνο αν αφήσουμε την ε, ε, Τελείωσε αρρύθμιση την εκμετάλλευση των δασών. Θα πρέπει λοιπόν να ε, εμποδιστεί η υπερεκμετάλλευση των δασών. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολύ σημαντική λοιπόν, έχει πολύ σημαντικό ρόλο να επιτρέψει τη διαφοροποίηση των οικονομιών αυτών των χωρών καθώς και να ρυθμίσει ένα περιορισμένο ε, ποσοστό εξαγωγών προς τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Ευχαριστώ κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα της ε, ξυλίας των δασών θα μας απασχολήσει και στο μέλλον ασφαλώς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δοθεί παράλληλα αυτές τις συμφωνίες και υποστήριξη ενίσχυση για την έρευνα. Και ιδιαίτερα να μεριμνήσουμε ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Καμερούν και το Κόγκο να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτυχθούν περισσότερο κατά τρόπο και οικολογικό και βιώσιμο. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα έτσι ώστε να προστατεύσουμε το μέλλον του ξύλου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 40% της έκτασης του Καμερούν το καλύπτουν τα δάση ακόμη, πρέπει να πω. Ωστόσο, το Καμερούν είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ξυλίας ε, της Αφρικής και παρουσιάζει μαζική αποψήλωση δασών έχουν χαθεί τα τελευταία 15 χρόνια τεράστιες εκτάσεις ε, ξυλίας και πολύτιμων ε, ειδών δέντρων από τη λεκάνη του ποταμού Κόγκο. Πρέπει λοιπόν ε, να αγωνιστούμε για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και ιδιαίτερα αυτούς τους ιδιώτες, τους ομίλους των ιδιωτών που εκμεταλλεύονται την γη κατά τρόπο μη βιώσιμο για να αποφύγουμε την πρώιμη αποψήλωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει λύσεις και σε σχέση με τα έσοδα που προέρχονται από την πόλη της Ξυλίας και οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν να λάβουν τις ευθύνες Ευχαριστώ. Επίτροπος τώρα παρακαλώ για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συζήτηση νομίζω ξεπέρασε το περιορισμένο πλαίσιο των εθελοντικών συμφωνίων εταιρικής σχέσης. Το δάσος δεν είναι μόνο πηγή ε, προϊόντος προς εμπορία, αλλά και πηγή ενέργειας και πηγή βιοπορισμού των πληθυσμών που ζουν κοντά σε αυτό και από αυτό. Ξέρω λοιπόν ότι η λύση δεν εξαντλείται, η λύση την οποία αναζητούμε δεν εξαντλείται με αυτές τις συμφωνίες. Είναι όμως ένα πρώτο σημαντικό βήμα πιστεύω. Και επίσης πρέπει να συζητήσουμε και με τις χώρες αυτές και να δούμε τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές. Ξέρουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι και οι χώρε αυτές έχουν άλλη ιστορία από τη δική μα. Εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους πριν από 50 χρόνια μόλις και μάλιστα σε συνθήκες πολύ δύσκολες και πολύ διαφορετικέ από αυτέ τις οποίες γνωρίσαν τα δικά μας κράτη στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Άρα έχουμε και να κάνουμε διαφθορά που πρέπει να καταπολεμηθεί και με εκμάθηση του τρόπου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Στην Αφρική ιδιαίτερα, αν κοιτάξτε, υπήρξε οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης. Άρα η Αφρική, τα αφρικανικά κράτη προχωρούν, προοδεύουν και βελτιώνονται. Ξέρω ότι μπορεί να φέρετε κάπως ζωφερή εικόνα αυτή τη στιγμή, αλλά η τάση είναι πάντως θετική. Εάν κάνουμε λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε αυτή την διαδικασία θα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή οι, αυτές οι συμφωνίες αυτό πράττουν ακριβώς με το Κονγκό, Μπραζαβίλ και το Καμερούν και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι επεξεργαζόμαστε αντίστοιχε συμφωνίες, μάλλον διαπραγματευόμαστε αντίστοιχε συμφωνίες και με την Ινδονησία οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα αλλά έχουμε βάσιμες ελπίδες. Ο κίνδυνος λοιπόν ε, είναι μηδαμινός εν προκειμένο γιατί πάνω απ' όλα στηριζόμαστε στη βούλησή μας και στην αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια θετική θεώρηση αυτής της υπόθεσης και ταυτόχρονα θα πρέπει να πιστέψουμε τις διαβεβαιώσεις του Κανκούν που προέκυψαν από το Κανκούν ότι και άλλες χώρες όσο από την Ευρώπη βλέπουν με αυστηρή ματιά το θέμα της διαφθοράς και θέλουν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους με αποφασιστικότητα. Αυτό βλέπουμε λοιπόν και ε, στην προκείμενη υπόθεση. Πολλά λοιπόν έχουμε να κερδίσουμε αυτές τις συμφωνίες. Και εν τέλει σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή και όχι μόνο το προσωπικό μου εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε και αντιπροσωπείε και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου και των κρατών μελών. Γι' αυτό είναι ένα από τα μελήματα που είναι κοινά μεταξύ Επιτροπή και κρατών μελών. Η δουλειά δεν είναι μόνο δηλαδή τη Επιτροπή. Σε πολλέ περιπτώσει, ιδιαίτερα η παρουσία και η συνδρομή των κρατών μελών ήταν πολύτιμη για να προχωρήσουμε σε αυτήν την υπόθεση. Θα παρακολουθούμε λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην εποπτεία. Είναι μια διαδικασία υγιής, μια διαδικασία η οποία προχωρεί προς την ορθή κατεύθυνση και πιστεύω ότι εν τέλει θα δώσει τις απαντήσεις σε όλα τα στήματα που εθίγησαν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο εισηγητής κύριο Ζαντού. Ευχαριστώ Επίτροπε και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο και υπήρξε σε ευρεία συνένεση και ακριβώς σας υπενθυμίζω ότι μέσω αυτών των συμφωνιών ε, έχουμε μια πολιτική υποφορά και την ε, κοινωνία των πολιτών και το περιβάλλον και την οικονομία οπότε πρόκειται με αυτόν τον λόγο για έναν μοχλό για βιώσιμη ανάπτυξη στις αφρικανικές χώρες και αυτό είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές. Το βασικό ίσως το μόνο στοιχείο δημοκρατικότητας είναι η ψήφος στις προεδρικές εκλογές είδατε τι έγινε με την ακτή Λεβαντοστού αλλά επομένω αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ενισχυθεί η των πολιτών, να συμμετέχει με πάγιο τρόπο σε ε, εφαρμογή τέτοιων συνθήκων ε, όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας, την εκμετάλλευση των δασών, όσον αφορά την κατανομή των σχετικών εισοδημάτων, που τα είπαμε και χθε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένω, νομίζω ότι μόνο με τέτοιου είδου αναβάθμιση τη κοινωνία μπορεί κανεί να απαντήσει στο αντεπιχείρημα που αφορά το τι γίνεται με την Κίνα και γιατί εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μια στενή συνεργασία με τα ισχυρά μας ε, ε, κριτήρια ε, μας λένε αυτές οι χώρες το θέλουν τα κριτήρια τελικά στα αυστηρά ενώ η Κίνα μας δίνει εύκολα κριτήρια που δίνουν στη λαϊλασία του περιφάροντος και επομένως το σύστημα το οποίο υπάρχει ο κίνδυνος να επιβάλλει η Κίνα αυτό θα συνεπιφέρει όμως η Ευρώπη είναι μια μεγάλη αγορά για το τροπικά δάση. Όμως και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλους ότι πρόκειται για σταθερή αγορά, αγορά που ξέρει να πληρώνει και αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα, ως υπομόχλιο στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστούμε που συνεργαστήκατε με το Κοινοβούλιο. Ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία μας μαζί σας. Uh, Σας ευχαριστούμε. Η κοινή συζήτηση εδώ τελειώνει γιατί έχουμε και μια πρόταση για ψήφισμα ούτω ώστε να ολοκληρωθεί και είναι συζήτηση. Η δε ψήφο θα γίνει στι 12.30 την Τετάρτη. Το επόμενο θέμα τώρα όμω για την κοινή συζήτηση